αυτά του κάθε Προέδρου της συνεδρίας, αλλά το βασικό φάρμακο είναι να ψηφίσουμε, ψηφίζουμε λιγότερα κείμενα και να τα ψηφίζουμε καλύτερα. Πρόεδρος, λοιπόν, πρώτον, αν μερολήπτησα θα ήμουν ευγνώμων να μου το λέγατε που μερολήπτησα και δεν ήμουν ουδέτερος θα ήμουν πρόθυμος να συζητήσω μαζί σας το θέμα. Όμως αντέδρασα αλλεργικά επειδή ακούστηκαν κάποια λόγια το ότι είναι λοιπόν έσχος δικό μου, ότι όλα αυτά είναι ανόητα, ότι επελέγει μια γλώσσα. Είναι μια γλώσσα που δεν είναι καθόλου ευγενική και κοινοβουλευτική στον τόνο της και γι' αυτό ενοχλήθηκα. Κατά τα άλλα προηγούμενα στο παρελθόν είχαμε περισσότερο χρόνο και για τις παρεμβάσεις και για τις ψηφοφορίες. Είχαμε ολομέλειες και την Παρασκευή το πρωί που εργαζόμασταν τότε. Μπορεί κανείς να λέει να έχουμε περισσότερο χρόνο για τις παρεμβάσεις. Από την άλλη πλευρά όμως ε, όλα στριμώχνονται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε πολύ λίγο χρόνο. Κατά τα άλλα θα πρέπει να επισημάνω ότι στις Βρυξέλλες ψηφίζουμε λιγότερο από ότι στο Στρασβούργο. Θα ήθελα να δώσουμε τις ευκαιρίες στους συναδέλφους τώρα να κάνουν τις επεξηγήσεις ψήφους, του. ψήφους των. Παρακαλώ. Καταρχήν όσον αφορά την έκθεση Φερνάντες ε,